Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, θεωρούνται δεκτά. Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας <clears throat> πέστηλαν στον Πρόεδρο δύο αιτήματα άρσης κοινοβουλευτικής ασυλίας για τους κυρίους κυρίους Γιάλκ και δύο επίσης ε, αιτήματα άρσης ε, για τον κύριο Λεπένα στα πλαίσια δικαστικών ε, διαδικασιών σύμφωνα με τον κανονισμό τα αιτήματα αυτά παραπέμπονται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Έλαβα επίσης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα